Καλημέρα σας. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Είχα ένα πρόβλημα. Θέλω να σας υπενθυμίσω κάτι το οποίο ξέρετε ήδη. I want to inform also that in this afternoon... Σήμερα το απόγευμα θα ξεκινήσουμε με την γνωμοδότηση για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πλοήγησης με δορυφόρο και μετά θα συνεχίσουμε με την Ασφάλεια και στη συνέχεια θα έχουμε συνεδρίαση του Διευρυμένου Προεδρίου. Αν δεν έχετε άλλες παρατηρήσεις, θεωρώ ότι έχει εγκριθεί η ημερησία διάταξη και μπορούμε να προχωρήσουμε. Αλλά έχω και κάποιες ανακοινώσεις ως Πρόεδρος. 8 Μαΐου θα λάβει χώρα μια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας από τις 11.30 ως 12.30 με στόχο να συζητήσουμε ένα σχέδιο ψηφίσματος που έχει προετοιμαστεί από την κυρία Γιατεμάκη για τις διαπραγματεύσεις για την ε, συνθήκη περί εμπορίου όπλων και η ίδια μέρα θα γίνει η συζήτηση μεταξύ 9.30 με 11.30 το πρωί για την ΕΦΙΑ άμυνα. Τα μέλη της Επιτροπής μας που θέλουν να παρακολουθήσουν αυτό το θέμα προσκαλούνται να είναι παρόντα. Και τώρα στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε σήμερα την πρώτη ανταλλαγή απόψεων με την για την εξέταση της γνωμοδότησης σε σχέση με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πλοήγησης με δορυφόρο, το Γαλιλαίο και το Έγνος. Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Τεχνολογίας και Έρευνας είναι επί της ύλης αρμόδια. Ο κύριος Τέρο είναι ο εισηγητής γνωμοδότησης από τη δική μας πλευρά. Σας δίνω μέσω στο λόγο κύριε Τέρχο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι θεωρώ ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι μια εξαιρετική πρόταση, πολύ ωφέλιμη, λαμβάνει υπόψη πολλούς τομείς των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας κτλ. Νομίζω ότι το δορυφορικό σύστημα πλοήγησης Γαλιλαίο και Έγνος δίδει στρατηγική ανεξαρτησία και στην Ένωση και στα κράτη-μέλη. Τα προγράμματα Γαλιλαίο και Έγνος είναι κοινοτικά προγράμματα, ε, θα έλεγα πρωτοπόρα και πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε πλήρως. Τα θέματα που έχουν σχέση με την άμυνα δεν περιλαμβάνονται πάρα πολύ ε, έντονα θα έλεγα στην πρόταση που επιμένει σε άλλους ομείς. Σε αυτή τη φάση, σαν παράδειγμα, δεν έχω πολλά να πω για τα θέματα τα δημοσιονομικά, αλλά το θέμα της ασφάλειας πρέπει να αντιμετωπιστεί σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Η συμπερίληψη των ωφελημάτων στον τομέα της άμυνας των δορυφορικών αυτών συστημάτων πλοήγησης έχουν υπογραμμιστεί στις εκθέσεις των αρμοδίων γενικών διευθύνσεων πέρυσι και οι άλλες υπερδυνάμεις δημιουργούν τα δικά τους συστήματα, τα δορυφορικά κυρίως γιατί τους διασφαλίζουν ασφάλεια και μετά χρησιμοποιούνται και για άλλους λόγους. Οι αμυντικές δυνατότητες και οι δυνατότητες στον τομέα της ασφάλειας έχουν αποδειχθεί σε πάρα πολλές ε, διεθνείς δράσεις, όπου στη Λιβύη, όπου ήταν περιορισμένες οι δυνατότητες τις οποίες είχαν ε, τα κράτη-μέλη. Το σύστημα Γαλιλαίου ήταν πολιτικό εξ αρχής και θα πρέπει να γίνεται αντικείμενο διαχείρισης επίσης από πολιτικές αρχές. Απ' την άλλη είναι ρεαλιστικό να παραδεχθεί κανείς ότι είναι διτής χρήσεως το πρόγραμμα αυτό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για λόγους ασφαλείας και στον πολιτικό τομέα και στον στρατιωτικό τομέα. Πρέπει να αναφερθούμε λοιπόν στα αμυντικά ωφέλη ε, προφανώς ανείχνευση, πλοήγηση, έρευνα, ε, διάσωση, ειρηνευτικές διαδικασίες και αύξηση της ανεξαρτησίας της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά θα πρέπει να τα υπογραμμίσουμε. Ένα τελευταίο σημείο ε, η εξάρτηση γενικά από τα αμερικάνικα συστήματα GPS ήταν ένα από τα επιχειρήματα που οδήγησαν στη δημιουργία του Γκαλιλαίου εξ αρχής. Σε εποχές ειρήνης η εξάρτηση αυτή δεν είναι κάτι το κρίσιμο, αλλά σε περιόδους ε, πολεμικών σειράξεων είναι σαφές ότι θα πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας αξιόπιστα συστήματα τα οποία να γίνονται αντικείμενο διαχείρισης από τους Ευρωπαίους. Γι' αυτό λοιπόν το σύστημα Γκαλιλαίο παρέχει προστιθέμενη αξία σε περιόδους κρίσης και γι' αυτό λοιπόν οι προτάσεις οι οποίες θα γίνουν έχουν μεγάλη σημασία. Κλείνοντας για το σύστημα Γκαλιλαίο υπάρχουν προφανείς πλευρές στον τομέα της άμυνας. Το πρόγραμμα αυτό θα κοστίσει περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ και περισσότερα από αυτά έχουν ήδη διατεθεί. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί και να εκμεταλλευτούμε το σύνολο των δυνατοτήτων του συστήματος και την προστιθέμενη αξία που παρέχει. Και αυτό περιλαμβάνει τις πλευρές της άμυνας και της ασφάλειας. Σε επίπεδο διαχειριστικό, διοικητικό, τα θέματα της ασφαλείας ανήκουν στο λεγόμενο δημόσιο ρυθμιστικό τομέα. Θα πρέπει τα ίδια τα κράτη-μέλη συνεπώς να αποφασίσουν εάν και πώς θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες στον τομέα της ασφαλείας του συστήματος. Κάποιες χώρες ίσως αποφασίσουν ότι δεν θα το κάνουν, κάποιες άλλες όμως έχουν πει ότι ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες του συστήματος. Θα τους δώσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές και τη δυνατότητα να το κάνουν. Είμαι δεκτικός στις ιδέες και στις προτάσεις των συναδέλφων στην πρόταση αυτή και θα ήθελα να σας καλέσω όλους να εκφραστείτε. Ευχαριστώ κύριε Τέρο για τη σύντομη παρέμβασή σας. Θα δώσω το λόγο εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον κύριο Φλαμπάν. Σας ευχαριστώ Κυρία Πρόεδρε, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να κάνω παρουσίαση της όλης πρότασης. Άλλωστε ο κύριο Στέρο πέρασε σε κάποια ουσιώδη λεπτομεριακά ζητήματα. Ουσιαστικά αναφερθήκατε εδώ πέρα σε μια διτή χρήση. Αυτό το οποίο θέλουμε εμείς να ευκρινίσουμε είναι ότι πέρυσι οι κανόνες πρόσβασης στην υπηρεσία GNSS και στην υπηρεσία PRS εγκρίθηκαν και προβλέπεται ότι κάθε κράτος μέλος θα μπορούσε να αποφασίσει από μόνο του με εντελώ κυρίαρχο τρόπο τον κατάλογο των χρηστών στους οποίους θα δώσει πρόσβαση στην παροχή της κρατικά ρυθμιζόμενης υπηρεσίας. Φέτος συνεργαζόμαστε προκειμένου να καταλήξουμε σε κάποια ελάχιστα κοινά πρότυπα τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζουν όλα τα κράτη-μέλη τα οποία θέλουν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία PRS. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύουμε ότι η χρήση της υπηρεσίας PRS θα πλησιώνει ουσιαστικά από όλα αυτά τα νομοθετικά κείμενα. Αυτή είναι η απάντηση που έχω να δώσω στις παρατηρήσεις που έκανε ο κύριος Στέρο. Σας ευχαριστούμε για τις παρατηρήσεις σας. Δίνω το λόγο στην κυρία Κοπά. Είναι η πρώτη στο κατάλογο μιλητών. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το σχέδιο αυτό κανονισμού είναι μια τροποποίηση του κανονισμού 2008 για την ε, ρύθμιση των προγραμμάτων Γαλιλαίος και Άγνος. Θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να πούμε ως μέλη της Επιτροπής μας για τα θέματα αυτά. Σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση. Εμείς είναι φυσικά θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα του ελέγχου από την πλευρά του Κοινοβουλίου και να εξασφαλίσουμε μια ε, ορθή δημοσιονομική διαχείριση. Και γι' αυτό η γνωμοδότησή μας τονίζει το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να τύχει τακτικής ε, πληροφόρησης για την εφαρμογή του προγράμματος αυτού, αλλά έχει και κάποιες αμβολίες για το ότι η διατύπωση του άρθρου 32 είναι η καλύτερη. Εγώ δεν είμαι εμπειρογνώμων για τα θέματα του προπολογισμού, αλλά είχα την εντύπωση ότι δίδονται υπερβολικέ εξουσίε στην Κομισιόν βάσει του κανονισμού αυτού. Η Κομισιόν έχει την ευθύνη του να εξασφαλίσει τα οικονομικά συμφέροντα τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει το δικαίωμα να κάνει λογιστικό έλεγχο των ε, αντισυμβαλόμενων και ε, δικαιούχων μαζί με το ελεκτικό συνέδριο. Αλλά ποιο θα ελέγξει την ίδια την Κομισιόν. Ίσως χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο για να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα δημοκρατικού ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να έχουμε την ευκαιρία με την ενδιάμεση αναθεώρηση να μπορεί η Κομισιόν να μα δώσει περισσότερε πληροφορίε και στοιχεία για τη δημοσιονομική διαχείριση. Αυτό είναι ένα γενικό σημείο σε σχέση με τα ειδικά θέματα τη επιτροπή μα. Νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσετε τη σημασία αυτού του συστήματος για την ανεξαρτησία και την ε, αυτονομία της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και για δράσεις της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη και το ρόλο των τρίτων χώρων στο πρόγραμμα αυτό και να γνωρίσω την ανάγκη αιότητα της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα. Θα ήθελα όμως να θέσω και ορισμένα ερωτήματα προς την Κομισιόν. Πρώτον, με ποιο τρόπο εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία των ευρωπαϊκών συστημάτων όταν χρειαζόμαστε χρηματοδοτική και τεχνική αρρωγή από τρίτες χώρε Δεύτερον, επειδή θεωρώ ότι αυτό θα είναι θέμα που θα αντιμετωπιστεί με μια συμφωνία συνεργασία βάσει του άρθρου 28 του κανονισμού, πώ θα εξασφαλίσουμε ότι οι τρίτε χώρε δεν θα χρησιμοποιήσουν αυτό το σύστημα για στρατιωτικού λόγους, όπως παραδείγματο χάρη για την κατεύθυνση βαλιστικών πυράβλων. Τρίτον, θα ήθελα να γνωρίζω αν ανοίγουμε αυτή τη δυνατότητα σε όλες τις χώρες ή αν θα έχουμε πρόσθετα κριτήρια, όπως παραδείγματος χάρη η υποχρέωση για την αρμόδια χώρα να έχει συνάψει μια συμφωνία ασφάλειας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, σε σχέση με την προστασία κρίσιμων υποδομών, ο προπολογισμό ο οποίος προτείνει καλύπτει όλο το κόστος ή εναπόκειται στα κρατημέλη που υποδέχονται αυτές τις υποδομές να το πράξουν αυτό. Και εδώ υπάρχει και το θέμα της εφαρμογής κοινή δράσης του Συμβουλίου του 2004. Θα ήθελα να καλωσορίσω την μνήα στην εισαγωγή της ανάγκης να υπάρξει μια επικαιροποίηση αυτής της απόφασης. Θέλω να σας πενθυμίσω ότι ήταν η δική μας Επιτροπή που υπογράμμισε την ανάγκη να είναι πιο προληπτικού χαρακτήρα οι πρόνοιες αυτού του νομοθετήματος και θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αναθεώρησης. Τέλος, χαιρετίζω την προσθήκη της ανάγκης να υπάρξει συνεργασία ε, μεταξύ Κομισιών και Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σε ό,τι αφορά σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια της Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Λόιζινγκ έχει το λόγο. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω στα γερμανικά. Εγώ μπορώ να συμφωνήσω με πολλά από αυτά που είπε η προλαλή σας ομιλήτρια και επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Τέρχο για τις ε, δηλώσεις του. Σε ορισμένα σημεία με ε, χαροποιεί γιατί ξέρω ότι έχει τονιστεί ίσως υπερβολικά η στρατιωτική διάσταση του Γαλιλαίου και χαίρομαι όταν υπάρχει και η δήλωση από μέλη της Επιτροπής μας που να καταδεικνύουν ότι υπάρχει ακριβώς αυτός ο στρατιωτικός δυνητικά χαρακτήρας στο Γαλιλαίο. Εγώ θέλω να περιοριστώ στα θέματα προϋπολογισμού. Όταν έχουμε ένα σχέδιο το οποίο έχει τόσο ευρεία δυνατότητα εφαρμογή σε στρατιωτικό επίπεδο, πρέπει να μιλήσουμε για διτή χρήση ή ακόμα και για ένα πρόγραμμα το οποίο είναι σχεδόν αποκλειστικά στρατιωτικού χαρακτήρα. Αλλά θα πρέπει να θέσουμε και το θέμα της διαφάνειας σε επίπεδο προϋπολογισμού. Βάσει των ε, ερευνών μου, περίπου 1,7 με 2 δισεκατομμύρια ε, θα πρέπει να προσθεθούν στο σχέδιο αυτό και θα ήθελα να ξέρω από πού θα προέλθουν τα χρήματα αυτά. Και θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο αυτή η κατά κύριο λόγο στρατιωτική ε, χρήση του Γαλιλαίου οδήγησε στο ότι οι Κινέζοι δεν μπορούν πια να συμμετέχουν σε αυτό το σχέδιο. Στο παρελθόν υποτίθεται θα ήταν ένα κοινό εγχείρημα μαζί με την Κίνα και αυτό θα μπορούσε να ελαφρώσει τη συνεισφορά του Ευρωπαίου φορολογούμενου, ιδίως σε μια εποχή έντονης οικονομικής κρίσης. Όταν λοιπόν έχουμε ένα σχέδιο το οποίο έχει κυρίως στρατιωτική ε, λειτουργία, κατά την δική μου άποψη δεν θα έπρεπε να χρηματοδοτείται από μη στρατιωτικό προϋπολογισμό όπως αυτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα ήθελα επίσης να τονίσω την ανάγκη να υπάρξει απόλυτη σαφήνεια σε σχέση με τη διαφάνεια του προϋπολογισμού, τι χρηματοδοτείται, από ποια θέση του προϋπολογισμού και για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται το κάθε κονδύλιο. Ευχαριστώ. Κύριος ε, Τσάμπολ. Um, um, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Δεν είμαι εμπειρογνώμων σε ζητήματα Γκαλιλαίο, αλλά το πραγματικό κόστος δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Δεν έχει δοθεί ακόμα ο πλήρης προπολογισμός. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή προβλέπει ένας προπολογισμός για την τρέχουσα εργασία και δημιουργία του συστήματος αυτού. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, δεν είμαι ειδικό στο ζήτημα, αυτό μου έχουν πει πάντως, πρώτον αυτόν. Δεύτερον, αν δεν γνωρίζουμε το τελικό κόστος, το συνολικό κόστος, ο συναδελφό μου αναφέρθηκε στη στρατηγική ανεξαρτησία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι ουσιαστικά είναι το βασικό πλεονέκτημα, το βασικό θετικό στοιχείο του συστήματο. Με ποιο τίμημα όμω πετυχαίνουμε το θετικό αυτό χαρακτηριστικό. Αν δεν γνωρίζουμε το συνολικό κόστο ή το κόστο του καλλιλέου αυτή τη στιγμή και πόσο κοστίζει για μη στρατιωτική χρήση, τότε ποιο θα είναι το επιπλέον κόστο τη διτή χρήση. Μήπω καταλήξουμε με ένα τεράστιο επιπλέον ποσό. Η εντύπωσή μου λοιπόν είναι ότι ε, αν δεν γνωρίζουμε ακριβώς το κόστος τόσο για την στρατιωτική και τη μη στρατιωτική χρήση και το τι κερδίζουμε τελικά με την περίφημη αυτή στρατηγική ανεξαρτησία, αν δεν αποδεχθεί αυτό το πράγμα, τότε δεν θα είμαι σε θέση να υποστηρίξω το εγχείρημα αυτό. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γκάλερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχήν, πιστεύω ότι τα τεχνολογικά πρότυπα του Γαλιλαίου και του Έγνος μας επιτρέπουν χρησιμοποιήσει και για πολιτικούς και για στρατιωτικούς σκοπούς. Το γεγονός ότι οι Κινέζοι έχουν αποσυρθεί από το πρόγραμμα αυτό μπορεί να είναι προς όφελός μας. Γιατί φοβόμουν ότι οι Κινέζοι θα κάνανε αυτό το οποίο κάνουν πάντα ότι ουσιαστικά θέλουν να αντιγράψουν και να χρησιμοποιήσουν για δικούς τους στόχους την τεχνολογία και την τεχνογνωσία ενό τέτοιου προγράμματο. Λοιπόν, το να αφήσουμε ένα τόσο προηγμένο τεχνολογικό πρόγραμμα να αντιγραφεί από του Κινέζου, αυτό δεν θα ήταν πολύ καλή ιδέα και να έχουμε τον ανταγωνισμό του. Δεν θα θέλαμε λοιπόν να χρησιμοποιηθεί για άλλου στόχου αυτή η τεχνολογία. Κατά τα άλλα, θεωρώ ότι, όπως είπε και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, όταν θέλουν τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν και για στρατιωτικούς στόχους αυτό το σύστημα, μπορούν να το κάνουν. Αλλά αυτό δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια αυτόνομη απόφαση που λαμβάνεται από τα κράτη-μέλη, αυτά τα οποία κάνουμε από κοινού ως Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απόλυτα λογικό να τα κάνουμε από κοινού μια πολιτική διαστήματος παραδείγματος χάρη, η οποία θα μπορέσει να εξασφαλίσει και την πολιτική μας ασφάλειας και την ε, πολιτική ασφάλειά μας. Αν θέλουμε να έχουμε παραδείγματος χάρη μια στρατιωτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να έχουμε και τις απαραίτητες τεχνολογίες να εξασφαλίσουμε την ε, αποτελεσματική στήριξη μιας τέτοιας αποστολής. Δεν θέλουμε να έχουμε σπατάλη πόρων και ικανοτήτων σε αυτές τις ε, αποστολές και με τον τρόπο αυτό να σωρεύεται το κόστος των δράσεών μας. Πιστεύω ότι ο έγνος είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα αν το συγκρίνουμε με το αμερικάνικο σύστημα GPS, ότι είναι πολύ πιο επακριβές το σύστημα έγνωση. Γιατί το GPS όμως δεν έχει τόσο μεγάλη ακρίβεια, γιατί οι Αμερικανοί έχουν κρατήσει μόνο την τεχνολογία, την τεχνολογία ακριβίας μόνο για το στρατιωτικό τομέα και μας δίνουν ασαφέστερες συντεταγμένες για την πολιτική χρήση. Ενώ εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την πλήρη ακρίβεια του έγνος και για πολιτικές αποστολές. Δεν αποκλείται λοιπόν μια τέτοια δυνατότητα. Θα ήθελα εδώ να μου διευκρινίσει καλύτερα η Κομισιόν πώς θα μπορούσε το έγνος και το Γαλιλαίος να χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν τις ε, μικτές στρατιωτικές και πολιτικές αποστολές στα πλαίσια της ΚΕΠΑ και πώς συνδέονται με την συμφωνία μεταξύ ΕΖΑ, ΕΝΤΑ και Κομισιόν για την έρευνα στον ε, τομέα της ασφάλειας και ακριβώς αυτό όπως ανέφερα πώς θα μπορέσουν με τον τρόπο αυτό να ενισχύσουν περισσότερο τις αποστολές της ΚΕΠΑ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα στα πλαίσια της συζήτησης να θέσω ορισμένες ερωτήσεις. Διάβασα με πολύ ενδιαφέρον το έγγραφο το οποίο λάβαμε για τη σημερινή συνεδρίαση. Πράγματι είναι πληρέστατο και ενδιαφέρον. Σήμερα αναφερόμαστε σε σχέδια, σε προγράμματα μάλλον, τα οποία ανήκουν στα πλέον σημαντικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν στεφθεί από επιτυχία η ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού, και το ελπίζουμε όλοι, θα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία της Ένωσης. Αν αποτύχει όμως, αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε θέση να ξεκινήσει μακροπρόθεσμα προγράμματα με ουσιαστικά τεχνολογικά βήματα. Το σύστημα αυτό πρέπει να είναι λειτουργικό το 2020 μέχρι τότε. Θα πρέπει να ξοδέψουμε ακόμα 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα ερωτήματα που τίθενται είναι τα εξής. Λοιπόν, μέχρι τώρα περνάγαμε σε συγκεκριμένες φάσεις. Υπήρχε η φάση σχεδιασμού, και σήμερα βρισκόμαστε στα θέματα της λειτουργίας του συστήματος και ε, στρέφουμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς θα γίνουν τα πράγματα πρακτικά, ποια είναι τα στοιχεία του συστήματος τα οποία έχουν ήδη δημιουργηθεί και τοποθετηθεί. Η δεύτερη ερώτηση αφορά τις στρατιωτικές δυνατότητες τις οποίες παρέχει το σύστημα αυτό γνωρίζουμε ότι οι περισσότερες χώρες που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι παράλληλα και μέλη του ΝΑΤΟ. Διαρωτώμε λοιπόν τι θα γίνει με τους ενόπλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν η χώρα τους ανήκει στην Ένωση αλλά ανήκει και στο ΝΑΤΟ διότι ξέρουμε ότι στο ΝΑΤΟ επικρατεί η τεχνογνωσία και η τεχνολογία η Αμερικανική. Η τελευταία ερώτησή μου αφορά τους τόπους εργασίας. Μου λέγουν ότι το σύστημα αυτό θα επιτρέψει στην Ευρώπη τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε διάφορες περιφέρειες και μάλιστα ιδιαίτερα επί υψηλού επίπεδου τεχνολογικά θέσεις εργασίας. Συμφωνούμε. Διαβάζοντας τα έγγραφα όμως, εγώ δεν βρήκα καμία πληροφορία για την κλίμακα δημιουργίας. Μιλάμε για χίλιες θέσεις, δυο χιλιάδες, πέντε χιλιάδες, πόσες. Και ο Κάνει κανείς κάποιες σκέψεις διαβάζοντας τις προτάσεις αυτές βλέπει ότι έγινε και έρευνα από το 2007 μέχρι το 2009 και στην κοινή γνώμη. Αυτά είναι λίγο πριν από τις εποχές λιτότητας. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει κάπως πιο νοπές εντυπώσεις για την αντίδραση του κοινού στο πρόγραμμα. Ευχαριστώ λοιπόν. Πριν δώσω το λόγο στην Επιτροπή για να απαντήσει στις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Έχω την αίσθηση ότι το πρόγραμμα αυτό είναι ένα στρατηγικής φύσης πρόγραμμα. Αν πράγματι πετύχουμε εδώ, τότε θα αποτελέσει σαφώς τμήμα της πολιτικής συνοχής, της πολιτικής ΚΕΠΑ και όχι μόνο εξοικονομεί χρήματα, αλλά έχει σημασία να χρηματοδοτήσουμε ό,τι απομένει για να πετύχουμε έτσι και άλλους στρατηγικούς στόχους. Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν είναι πολύ εύκολο να απαντήσω σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Καλύψανε πάρα πολλούς τομείς οι ομιλητές. Θα προσπαθήσω παρόλα αυτά να είμαι σύντομος και να καλύψω όλες τις παρατηρήσεις. Καταρχάς, πού βρισκόμαστε σήμερα με το πρόγραμμα αυτό άκουσα κάποια αριθμητικά δεδομένα. Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι 5 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί μέχρι στιγμής για το σύστημα Γκαλιλαίο. Με αυτά τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ τι έχουμε. Έχουμε δύο δορυφόρους οι οποίοι βρίσκονται σε τροχιά εδώ και κάποια χρόνια. Οι πειραματικοί λοιπόν αυτοί δορυφόροι μας δείχνουν ότι η ευρωπαϊκή τεχνολογία είναι σε θέση να παράγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία πετούνται στα πλαίσια του συστήματος Γκαλιλαίου. Δεύτερον, έχουμε δύο επιχειρησιακούς δορυφόρους, εκτοξεύθηκαν στις 21 Οκτωβρίου και δύο ακόμα επιχειρησιακοί δορυφόροι θα εκτοξευθούν φέτος. Στα πλαίσια των 5 δισεκατομμύριων ευρώ έχουμε κάποιες συμβάσεις με επιχειρήσεις προκειμένου να κατασκευάσουμε κάποιους δορυφόρους και προκειμένου να εξασφαλίσουμε την εκτόξευση δορυφόρων. Επίσης χρησιμοποιούμε όλη τη διαθέσιμη υποδομή τους, τα κέντρα εδάφους, καθώς επίσης και τα κέντρα εποπτείας, τα οποία έχουμε παντού στον κόσμο. Μέσα σε αυτά τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσαμε προκειμένου να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε μέχρι τα τέλη του 2015 μία συσώση στοιχεία δορυφόρων, 20 περίπου δορυφόρων. Αυτό θα κάνουμε με τα χρήματα που έχουμε μέχρι σήμερα. Χρειαζόμαστε όμως και απαραίτητα χρήματα προκειμένου να καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε το σύστημα 7 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Έχουμε καταλήξει στο ποσό αυτό το πολύ συγκεκριμένο, βασιζόμενοι στην εμπειρία που είχαμε από το παρελθόν, βάσει των συμβάσεων που ήδη ισχύουν και βέβαια συνεργαζόμαστε με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα διαστημικά συστήματα εδώ και 30 χρόνια και καταφέραμε να εξακριβώσουμε όλα αυτά τα αριθμητικά δεδομένα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών. Ξέρω ότι ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εθνικούς οργανισμούς διαστήματος, επομένως ελέγξαμε μαζί τους τα αριθμητικά αυτά δεδομένα του προπολογισμού. Αυτά λοιπόν για το τι έχουμε δαπανίσει μέχρι σήμερα και τι προβλέπουμε να κάνουμε με αυτά τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ έχουμε και το τέλος του σταδίου της ε, εγκατάστασης. Ε, πρέπει να ολοκληρωθεί η συνολική υποδομή, περιλαμβάνει 30 συνολικά δορυφόρους και έχουμε βέβαια και τους απαραίτητους πόρους προκειμένου να καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε πλήρως και το σύστημα EGNOS, το οποίο ουσιαστικά βελτιώνει τις επιδόσεις του συστήματος GPS στην Ευρώπη. Όσον αφορά τώρα τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πώς γίνεται ο έλεγχος αυτός. Κοιτάξτε, ήδη υποβάλλονται πολλές αναφορές οι οποίες δείχνουν πώς προχωράει το πρόγραμμα. Κάνουμε επίσης πολύ συχνά σε τακτική βάση συναντήσεις με τα κράτη-μέλη μέσω του συστήματος επιτροπολογίας. Έχουμε μία επιτροπή προγράμματος όπου δείχνουμε στα κράτη-μέλη πώς προχωρούν τα πράγματα. Βέβαια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε φορά που το επιθυμεί έχει όλες τις απαραίτητες ε, αναφορές, εκθέσεις, ενδιάμεσες αναθεωρήσεις. Μπορούμε και στο κείμενο αυτό, αν θέλετε, να εντάξουμε όλες αυτές τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όσον αφορά τώρα τα ωφέλη. Σοβαρές ε, μελέτες ε, διενεργήθηκαν από τον οργανισμό του Ευρωπαϊκού GNSS, οι οποίες κατέδειξαν ότι μόνο και μόνο η εργασία μας στα πλαίσια της δορυφορικής ραδιοπλοήγησης μέσα στα επόμενα 20 χρόνια θα φτάσουμε σε ωφέλη της τάξης των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτές οι επενδύσεις είναι ιδιαίτερα αποδοτικές και ακόμα και αν δεν είναι πλήρως επιχειρησιακό ακόμα το σύστημα, μπορούμε να πούμε ότι όλες αυτές οι εργασίες που γίναν τελευταία δέκα χρόνια από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μας έχουν επιτρέψει να φτάσουμε ένα υψηλότατο επίπεδο στα πλαίσια της ραδιοπλοήγησης και αυτή τη στιγμή για κάποιους πομπούς δέκτες χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Και αυτό έγινε χάρη σε επενδύσεις που έχουν γίνει στα πλαίσια του Γαλιλαίου και του Έγνος. Όσον αφορά τώρα τις ε, κοινέ δράσεις, υπάρχει μία μνήα στην πρόταση κανονισμού. Καταλαβαίνετε όμως ότι αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει αποκλειστικότητα της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γι' αυτό το λόγο ο Αντιπρόεδρος Νταγιάννη έστειλε μια επιστολή στην κυρία Άστον αναφερόμενο στην επικαιροποίηση αυτής της κοινή δράσης. Αναφέρθηκα έτσι αρκετά γρήγορα στις ερωτήσεις τις οποίες θέσατε. Τώρα, για το αν θα είναι το σύστημα αυτό διαθέσιμο σε τρίτες χώρες. Πρέπει να ξέρετε ότι τον Γαλιλαίο προσφέρει πέντε υπηρεσίες. Έχουμε ουσιαστικά την ανοιχτή υπηρεσία και την, και την υπηρεσία PRS. Όσον αφορά την, ανοιχτή, με συγχωρείτε, υπηρεσία, λειτουργούμε όπως το GPS, δηλαδή τα σήματα GPS διατίθενται δωρεάν για όλους τους χρήστες παντού στον κόσμο και αυτή η παροχή ανοιχτή υπηρεσίας θα εξακολουθήσει να ισχύει για όλους τους χρήστες παντού στον κόσμο. Όσον αφορά τώρα την κρατικά ρυθμιζόμενη υπηρεσία PRS, η υπηρεσία αυτή θα είναι διαθέσιμη για κάποιες τρίτες χώρες, αφού πρώτα όμως συνάψουμε συμφωνίες επίσημες με τις χώρες αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 218 της Συνθήκης. Ενδεχομένω να μην απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις, πάντως πιστεύω ότι κατά 80-90% έχω καλύψει τις παρατηρήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Όταν μιλάτε για το κόστος, μιλάτε για το κόστος των υποδομών. Γιατί για τις υποδομές είπα ότι έχουμε ήδη επενδύσει 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Χωρίς μικρόφωνο μιλητής ο κύριος Κάμπελ. Το κόστος λοιπόν που εντοπίζεται εδώ τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ για την 7 ετία 2014-2020 δεν σημαίνει ότι μετά από το 2020 δεν θα υπάρχει κόστος υποδομής γιατί από τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί μια υποδομή θα πρέπει να την κρατήσουμε σε λειτουργία, να την βελτιώνουμε, να την επικαιροποιούμε, να ικανοποιούμε τις ανάγκες των χρηστών. Ναι, η δημόσια αυτή υπηρεσία που είναι η πλοήγηση με δορυφόρο θα εξακολουθήσει να χρειάζεται χρηματοδότηση απλώς και μόνο για την συντήρηση του συστήματος. Είναι γεγονός τώρα ότι παραλλήλως Προσπαθούμε να έχουμε και έσοδα από ορισμένε υπηρεσίε του Γαλιλαίου. Από τι πέντε υπηρεσίε Γαλιλαίου, μία είναι η λεγόμενη εμπορική υπηρεσία και οι μελέτες δείχνουν ότι τουλάχιστον μέσα στα πρώτα χρόνια λειτουργία, τα έσοδα αυτής της εμπορικής ε, υπηρεσίας δεν θα επαρκέσουν για να καλύψουν το κόστο τη λειτουργία του συστήματο. Εντάξει, λέει η πρόεδρο. Ένα ακόμα ερώτημα. Ευχαριστώ. Ίσως είναι θέμα αγνιάς μου για το ζήτημα αυτό που θέτω το ερώτημα αυτό. Αλλά είπατε ότι ο Γαλιλαίος θα προσπαθήσει να είναι και κερδοφόρος. Δηλαδή θα γίνει μια εμπορική υπηρεσία σε κάποια χρονική στιγμή. Έχετε κάποια στοιχεία, κάποια ανάλυση που δείχνει κατά πόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα μέχρι τώρα έχει χρηματοδοτηθεί μόνο από δημόσια ταμεία. Δεν θα μας πάει κανείς στο πάνελ του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για το θέμα αυτό, ιδίω εφόσον πρόκειται για χρηματοδότηση μόνο από δημόσια κονδύλια. Ναι, να απαντήσετε αν θέλετε, η Κομισιόν και πάλι. σε ό,τι αφορά την εμπορική υπηρεσία. Ναι, πράγματι. Σα είπα ότι από τι πέντε υπηρεσίε του Γαλλίου μία έχει εμπορικό χαρακτήρα και οι μελέτες έδειξαν σε 15 χρόνια αυτή η υπηρεσία θα πρέπει να καλύπτει το 1 δέκατο του κόστους λειτουργίας του συστήματος. Αλλά κανείς δεν θεωρεί ότι θα μας φέρουν ενώπιον του πάνελ του ΠΟΕ για το θέμα αυτό, γιατί δεν υπάρχει θέμα ανταγωνισμού σε σχέση με τα ζητήματα αυτά. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να θέσουμε στη διάθεση ορισμένων εμπορικών φορέων τις ικανότητες του συστήματος Γαλιλαίου βεβαίως και για να το επιτύχουμε αυτό θα πρέπει να έχουμε και κάποια συνεισφορά αυτών των φορέων για την υλοποίηση αυτού του συστήματος και θα έχουμε λοιπόν αυτά τα έσοδα τα οποία θα καλύπτουν το 1 δέκατο του κόστου λειτουργίας του συστήματος. Ευχαριστώ, ελπίζω ότι σας ικανοποίησαν οι ερωτήσεις. Δίνω το λόγο στον εισηγητή για να κλείσει τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Θα συνεχιστεί η συνεργασία με τους κοιόδης συγγητές και ελπίζω να βρούμε μια σωστή λύση. Okay. Καλώς λοιπόν. you have an intervention? Κύριε Γκάλερ, κάτι θέλετε να πείτε. Ίσως να το πω αγγλικά για να με καταλάβετε καλύτερα. Θα ήθελα μια διευκρίνηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον τρόπο με τον οποίο τον Καλλιλέο και Έγνος μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα για να υποστηριχθούν καλύτερα οι δράσεις μας στον τομέα της άμυνας, της ασφάλειας και γενικότερα οι εξωτερικές δράσεις μας. Έχετε κάποιες ιδέες πιο συγκεκριμένες. Άλλη μία ερώτηση λοιπόν. Μία ακόμα ερώτηση και μετά θα δώσετε κοινή απάντηση. Κύριος Λάντσμπεργκης. Πώς συνδέεται η διαδικασία αυτή για τον Καριλαίο και πώς συνδυάζει μάλλον την πολιτική και τη στρατιωτική χρήση του διαστήματος καμία μα καμία αναφορά στο ΝΑΤΟ. Αγνοείται το ΝΑΤΟ εντελώς. Τι σημαίνει αυτό, τι είναι αυτό. Αναφέρεστε για τον συντονισμό σε τεχνικές πλευρές, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, αλλά υπάρχει και το ΝΑΤΟ. Μεγάλη υπηρεσία. Προφανώς και θα πρέπει να συντονιστούμε με τον ΝΑΤΟ. Ή θα πρέπει επίσης και να κάνουμε ότι δεν υπάρχει το ΝΑΤΟ, να το αγνοήσουμε πλήρως. Κοιτάξτε, υπάρχει πολύ ενδιαφέρον όπως βλέπετε για το θέμα στην Επιτροπή μας. Έχετε τον λόγο για να απαντήσετε στις δύο τελευταίες ερωτήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σχετικά με τη χρήση από το ΝΑΤΟ, η πρόταση κανονισμού μας είναι μια πρόταση η οποία αναφέρεται στα της διαχείρισης και στον προϋπολογισμό. Δεν περνάμε εμείς τις λεπτομέρειες της χρήσης των πέντε επιρρησεών. Σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης από τον ΝΑΤΟ θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ήδη πέρυσι έγινε δεκτός ένας κανονισμός που ονομάζεται «Κανόνες πρόσβασης στο σύστημα PRS» και στα πλαίσια αυτών των κανόνων λέγουμε ότι τρίτες χώρες, Νορβηγία, Ελβετία κυρίως, αλλά και διεθνείς οργανώσεις πιθανώς στο ΝΑΤΟ, μπορεί να έχουν ε, πρόσβαση στο PRS ανάλογα με την υπογραφή μιας συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο 218 της Συνθήκης. Γύρω τώρα από την χρήση του συστήματος από το Συμβούλιο ή τον παλαιό λεγόμενο δεύτερο πυλώνα. Αυτό δεν το αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες συνθήκες έτσι ώστε να μπορεί να υπάρξει χρήση του συστήματος από κάθε χρήστη στις βέλτιστες δυνατές συνθήκες κάτω από ειδικέ περιπτώσεις. Αλλά τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα για την χρήση του συστήματος PRS στα πλαίσια συγκεκριμένων δράσεων του τέος στο δεύτερο πυλώνα. Thank you. Ευχαριστώ. Αν δεν έχουμε άλλο ερώτημα. Μπορείτε να συνεχίσετε ε, διμερώς τις συζητήσεις αυτές. Το θέμα αυτό έχει κλείσει και προχωρούμε στο επόμενο θέμα στην ημερησία διαταξή μας. Το 2011, το Δεκέμβριο, πήραμε το δικαίωμα να, προ... να προετοιμάσουμε περισσότερες εκθέσεις πρωτοβουλίες, μία από τις οποίες είναι η έκθεση για την κυβερνοασφάλεια και κυβερνοάμυνα. Ο εισηγητής μας είναι ο κύριος Κέλαμ αλλά η σημερινή μας συνάντηση δεν αφορά την έκθεση του κ. Κέλαμα, αλλά την πρόταση του Κομισιόν να δημιουργήσει ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Αντιμετώπισης του Κυβερνοεγκλήματος. Στο παρελθόν καλυπτόταν αυτό από ένα άλλο φορέα, την ΕΝΙΣΑ, και από το κέντρο αριστείας για την κυβερνοάμυνα της Ταλίνης. Σήμερα όμως έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με την Κομισιόν για την προστιθέμενη αξία που μπορεί να προσθεθεί, που να προκύψει από τη δημιουργία αυτού του νέου φορέα και σε σχέση με την δυνατότητα να δώσουμε μεγαλύτερη σύνοχη στις κοινέ μας πολιτικές στον τομέα αυτό. Θα δώσω λοιπόν το λόγο πρώτα στην Κομισιόν για το θέμα αυτό και στη συνέχεια εάν ο συνάδελφός μας ο κύριος Κέλλαμ θέλει να παρέμβει όπως και οι άλλοι συνάδελφοι θα τους δώσω τον λόγο. Η Κομισιόν λοιπόν έχει το λόγο για το θέμα αυτό της ασφάλειας. Ο εμπειρογνώμονας μας δεν έχει έρθει ακόμα. Προχωρήσετε τόσο γρήγορα με το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Κανονικά θα ερχόταν στις 4. Uh, Άρα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, αλλά με την σύμφωνη γνώμη του κυρίου Κέλαμ θα μπορούσε μάλλον να πάρει πρώτος αυτό το λόγο και στη συνέχεια να ακούσουμε και τον Δήμονα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Κέλαμ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε κάποιες νέες πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ε, ανάγκη για την ε, νέα αυτή πρωτοβουλία που υπάρχει για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για ζητήματα όπως η ασφάλεια των υποδομών και επίσης θα έχουμε και μια έκθεση όσον αφορά την ε, ε, νομική συνεργασία για διάφορα εγκλήματα, για διάφορες επιθέσεις σε κάποια συστήματα πληροφοριών. Η κυρία Κορτ θα επιληφθεί αυτού. Και έχουμε και την έκθεση για την ΕΝΙΣΑ. Η συγκεκριμένη πάντως έκθεση έχει να κάνει με τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο και ουσιαστικά θα πρέπει να βασίζεται στις κοινέ μας πολιτικές ε, άμυνας και ασφάλειας. Υπάρχει λοιπόν ένα ευρύ πλαίσιο το οποίο πρέπει να έχουμε κατά νου. Ποιους στόχους θέλουμε να επιτύχουμε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση, να υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική για την καταπολέμηση των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο. Θα πρέπει όλες οι πτυχές και διαστάσεις να συμπεριληφθούν. Θέλουμε επίσης μια συντονισμένη προσέγγιση, η οποία θα εντοπίζει τις βέλτιστες πρακτικές. Θέλουμε να γνωρίζουμε επίσης πώς μπορούν αυτές να εφαρμοστούν αποτελεσματικά. Και τίθεται επίσης και το ζήτημα του να μπορούμε να έχουμε μία θέση συντονιστή για την καταπολέμηση των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο. Αξίζει να κάνουμε κάτι τέτοιο, θα έχει νόημα να γίνει κάτι τέτοιο. Ποιε αρμοδιότητε θα έχει ο άνθρωπο που θα αναλάβει τη θέση αυτή. επίση πρέπει να ευθυγραμμίσουμε, να εξορθολογήσουμε την καταπολέμηση των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο στα πλαίσια της πολιτικής που ακολουθούμε για τις εξωτερικές υποθέσεις, για την άμυνα και την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιο ρόλο μπορεί να έχει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνα στα πλαίσια της κυβερνοασφάλειας και θα πρέπει επίσης να δούμε πώς μπορούμε να συλλέξουμε τις απαραίτητες πληροφορίες, πώς μπορούμε να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς μπορούμε να έχουμε επίσης καλή συνεργασία μεταξύ των εξωτερικών και εσωτερικών διαστάσεων της κυβερνοασφάλειας. Γιατί στην πράξη αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι δεν μπορεί κανείς να διαχωρίσει εύκολα τις δύο αυτές πτυχές, τις δύο αυτές διαστάσεις. Και βέβαια, θα πρέπει να ασχοληθούμε πολύ και με τις σχέσεις μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων. Θα πρέπει να αφαιρθούμε δηλαδή στις εταιρικέ σχέσεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα. Τις σχέσεις μας με τους εξωτερικούς φορείς, όπως για παράδειγμα το ΝΑΤΟ, το πώς μπορούμε να συγκεράσουμε τις αρμοδιότητές μας, πώς μπορούμε να κάνουμε καλύτερη κατανομή αρμοδιοτήτων και οι σχέσεις μας βέβαια με τις τρίτες χώρες και αυτές πρέπει να μας απασχολήσουν. Θα πρέπει να εμπλέξουμε και τις τρίτες χώρες. Και τίθεται βέβαια και το ζήτημα της ε, νομικής ευθύνης. Νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε για κάποια ελάχιστα νομικά πρότυπα. Και θα πρέπει να δούμε και τα πιο θετικά παραδείγματα που έχουμε και να δούμε επίσης τι θα γίνει με την σύμβαση αυτή την οποία δεν έχουν ακόμα υπογράψει, δεν έχουν επικυρώσει οκτώ κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε, να επικυρωποιήσουμε τη σύμβαση αυτή ή ουσιαστικά μπορούμε να συνεχίσουμε με την υφιστάμενη σύμβαση. και τίθεται και το ζήτημα της εξισορρόπησης ανάμεσα στην ελευθερία και την ευελιξία και τις κυρώσεις που θα πρέπει ενδεχομένω να επιβληθούν και τους περιορισμούς που θα πρέπει να υπάρχουν στην χρήση των συστημάτων πληροφοριών. Νομίζω ότι αυτά είναι τα σημαντικότερα ζητήματα τα οποία τίθενται και τα οποία θα πρέπει να διευθετηθούν στα πλαίσια της μελλοντική μας έκθεσης. Το εφιστάμενο χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής. Πρώτη εξέταση θα γίνει στην υποπιτροπή μας τον Ιούλιο, μέχρι τον Ιούλιο, δηλαδή πριν διακόψουμε για τις θερινές διακοπές. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών θα είναι στις αρχές περίπου Σεπτεμβρίου. Με απότερο στόχο να έχουμε μια δεύτερη εξέταση του σχεδίου έκθεσης μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου και έγκριση από την ΑΦΕΤ τον Οκτώβριο. Σας ευχαριστώ. Μπορούμε να συζητήσουμε πράγματι για αυτά που είπε ο κύριος Κέλα. Έχετε το λόγο, κύριε Κόπα. Θα ήθελα να παρέμβω για αυτά τα οποία για το έγγραφο της Κομισιόν. Μήπως πρέπει να περιμένουν να έρθει η Κομισιόν ή θέλετε να μιλήσω τώρα. Δεν είναι εδώ ο Ιδήμων, ο Επαΐων ίσως να περιμένουμε, να τον περιμένουμε. Γιατί μπορεί να είναι και άλλα τα ερωτήματα τα οποία θα τεθούν προς την Κομισιόν για να απαντήσει η Κομισιόν χωρίς να επαναλαμβανόμαστε. our... Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια τώρα για την έκθεση του κύριου Κέλαμ συγκεκριμένα. Κύριε Γκάλερ. Σας ευχαριστώ. Έχουμε τώρα το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές επιτροπές που ασχολούνται με το θέμα αυτό και από διαφορετικές οπτικές γωνίες για το ζήτημα αυτό της κυβερνοασφάλειας και νομίζω ότι είναι σωστό να το δούμε και στη δική μας υποεπιτροπή γιατί γνωρίζουμε ότι η πτυχή αυτή μας ε, εμπλέκει έμεσα ως Επιτροπή Ασφάλειας Νομίζω λοιπόν ότι είναι σαφές ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Είναι πολύ σωστό να συζητούμε για το θέμα αυτό. Το ερώτημα φυσικά το οποίο τίθεται σε σχέση με όλα αυτά είναι το εξής. Έχουμε διαφορετικούς φορείς οι οποίοι αντιμετωπίζουν την προστασία, την ε, ε, άμυνα από τις επιθέσεις στον κυβερνό χώρο. Όλα όμως αυτά Όλες αυτές οι ενέργειες γίνονται μέσα στον παγκοσμιστό, το World Wide Web. Υπάρχει μόνο ένας χώρος λοιπόν μέσα στον οποίο πρέπει να γίνεται αυτή η άμυνα, αλλά έχουμε πάρα πολλούς αμυντικούς φορείς ε, ούτως ποινή. με μεγάλη δυσκολία λοιπόν είναι το πώς θα βρούμε έναν τρόπο να συντονίσουμε τις διάφορες προσπάθειες, πώς θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα σύστημα το οποίο θα ξεπερνάει τα εθνικά σύνορα και τις εθνικές αρμόδιες αρχές και στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, στον ε, τομέα που επαφίεται και στρατιωτικών θεμάτων, θα είναι πολύ πιο ευαίσθητα τα θέματα αυτά, πολύ πιο ευαίσθητα από ότι σε άλλους χώρους άμυνας από το κυφερνό έγκλημα. γιατί φυσικά θα εμπλέκονται και ζητήματα βελτίωσης της ίδιας της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό πρέπει να είναι ένα πλήρες και συνολικό έργο και γι' αυτό ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτά τα οποία θα μας πει ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Ελπίζω λοιπόν ότι με αυτά που είπα κάπως γέμισα και τον κενό χρόνο, αλλά ίσως θα πρότεινα στο μέλλον όταν έχουμε μία συνεδρίαση στις 3 η ώρα και όταν το δεύτερο σημείο προβλέπεται να έρχεται το σημείο αυτό πρόκειται να είναι το δεύτερο σημείο. Ίσως ο εκπρόσωπος της Κομισιόν μπορεί να έρχεται και λίγο νωρίτερα. Και να παρακολουθεί και τη συζήτηση, ιδίως όταν έχουμε δύο θέματα όπως σήμερα, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους ως ε, αντικείμενο. Ίσως η Κομισιόν λοιπόν θα μπορούσε να λάβει υπόψη της για το μέλλον, όταν έχει να αντιμετωπιστεί ένα σύνολο από συναφή θέματα, θα είναι καλύτερο να υπάρχει ο εκπρόσωπος παρόν. Δεν μπορώ τώρα να πω τίποτα περισσότερο στον τομέα αυτό. Μπορούμε να κάνουμε ένα διάλειμμα βέβαια. Δεν φταίμε φυσικά εμείς αν η Κομισιόν δεν έχει στείλει τον εμπειρογνώμονά της για την... Αν μπορώ κυρία Πρόεδρε μπορούμε να στείλουμε ένα μήνυμα στην Κομισιόν ότι εφόσον δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για κάθε θέμα, θα ήταν σόφρον, όπως λέει και ο κύριο Γκάλερ, να είναι η εκπρόσωποι της Κομισιόν εδώ από την αρχή. Βεβαίω λέει η πρόεδρο. Γιατί ήδη έχει καθυστερήσει ο εκπρόσωπος. Μπορούμε να διακόψουμε για λίγα λεπτά γιατί είναι δύσκολο να μιλάμε για κάτι χωρίς την παρουσία της Κομισιόν, χωρίς συνομιλητή. Παρά το γεγονός ότι προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αν μπορεί κάποιος να προειδοποίησει τον ε, εκπρόσωπο της Κομισιόν, γιατί κλείσαμε το προηγούμενο θέμα τέσσερα λεπτά πριν από τις τέσσερις. Έχει χαθεί στο κυβερνόχωρο, λέει ο, ο αντιπρόεδρος, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, ίσως έπεσε θύμα εγκλήματος.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 Okay. Εντάξει, σας δίνουμε το λόγο για να μας παρουσιάσετε την πρωτοβουλία της Κομισιόν και θα υπάρξουν στη συνέχεια ερωτήσεις προς εσάς που θα πρέπει να είστε προετοιμασμένος να απαντήσετε. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. δεν ήταν κυβερνοεπίθεση, αλλά ήταν μια διακριτική μεταχείριση των ποδηλατών από τα άλλα θεσμικά όργανα. Εγώ δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω το χώρο σταθμεύσης ποδηλάτων στο Κοινοβούλιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την πρόσκληση προς τον εκπρόσωπο της Κομισιόν να σας πληροφορήσει για την πρόσφατη αυτή πρωτοβουλία για δημιουργία ενός κέντρου αντιμετώπισης του κυβερνοεγκλήματος Καταρχήν να σας παρουσιάσω το γενικό πλαίσιο. Ξέρετε λοιπόν πώς τα θέματα του κυβερνόχωρου και ιδίως τα θέματα κυβερνοεγκλήματος αποκτούν μεγαλύτερη σημασία στην πολιτική ατζέντα τα τελευταία χρόνια. Το 2010 είχαμε συμπεράσματα υπό Ισπανική Προεδρία για το κυβερνοέγκλημα και ένα από τα θέματα αυτά που ήταν στα συμπεράσματα του Συμβουλίου ήταν μια έκκληση από τα κράτη-μέλη προς την Κομισιόν να δημιουργήσει ένα κέντρο αντιμετώπισης του κυβερνοεγκλήματος και μέσα στην, ε, κυβε... στην κοινή στρατηγική για τα θέματα αυτά καθορίστηκαν πέντε κύριοι στόχοι για το κυβερνοέγκλημα μέσα στην πολιτική της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Κομισιόν έχει αναλάβει την υποχρέωση να δημιουργήσει αυτό το κέντρο. Για να καρποφορήσει τώρα αυτή η διαδικασία με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι καλά σχεδιασμένος, υπήρξε σε βάθος προπαρασκευαστική εργασία, <clears throat> μελέτες σκοπιμότητος, που έγινε από ένα εξωτερικό συνεργάτη. Είχαμε πολλές διαβουλεύσεις και με τους εμπλεκόμενους στα κράτη-μέλη για να μπορέσουμε <clears throat> να δούμε ποιες είναι οι ικανότητες που υπάρχουν για την αντιμετώπιση του κυβέρνου εγκλήματος και να δούμε πού θα μπορούσε να προκύψει προσθέμενη αξία για δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν πιο αποτελεσματική καταπολέμηση του κυβέρνου εγκλήματος. Στόχος μας ήταν λοιπόν να απαντήσουμε σε ερωτήματα όπως τι είδους λειτουργίες θα έπρεπε να έχει ένα τέτοιο κέντρο και επίσης πολύ σημαντικό πού θα έπρεπε να είναι αυτό το κέντρο. Είχαμε μια περιεκτική διαδικασία, υπήρξε διαβούλευση με τα κράτη-μέλη, με τους εμπειρογνώμονες, τους επαγγελματικούς κλάδους, φορείς όπως η ΕΝΙΣΑ. Και φαίνεται ότι όλο και περισσότερο συνειδητοποιούμε ότι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα του κυβερνοχώρου και του κυβερνοεγκλήματος πιο αποτελεσματικά, θα πρέπει να περάσουμε και πέρα από τα στεγανά τα οποία ισχύουν αυτή τη στιγμή στα κράτη-μέλη να βγούμε από χώρους οι οποίοι είναι και χωρισμένοι. Ο ένας είναι ο χώρος των αστυνομικών δυνάμεων, ο άλλος είναι του ιδιωτικού τομέα. Ο... Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη γνώση των ε, εμπειρογνωμόνων, είτε είναι δημόσιοι είτε είναι ιδιωτικοί, οι οποίοι εργάζονται για την ανθεκτικότητα των συστημάτων και του διαδικτύου. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν έχουν ληφθεί υπόψη στην προετοιμασία αυτής τη πρωτοβουλία. Στι 20 Μαρτίου η Κομισιόν ενέκρινε και μία ανακοίνωση για το θέμα αυτό και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για το γεγονός ότι είχε μόνο οκτώ σελίδες αυτή η ανακοίνωση. Προσπαθήσαμε λοιπόν να μην οδηγήσουμε σε θάνατο από ανία τον, ε, τους Ευρωπαίους πολίτες. Ε, δεν πρόκειται λοιπόν για μια γενικόλογη δήλωση, ούτε για μια ιδιαίτερα λεπτομερή έκθεση, αλλά η εστίαση του εγγράφου ήτανε ακριβώς για την δημιουργία ενός, ενός κέντρου για το κυβερνό χώρο και το κυβερνό έγκλημα. Αυτό το οποίο κάναμε ήταν καταρχήν να ε, απαριθμίσουμε τα είδη κυβερνοεγκλημάτων όπου θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει μια απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν τρεις ομάδες εγκλημάτων, καταρχήν τα κυβερνοεγκλήματα από οργανωμένες ομάδες, από ομάδες οργανωμένου εγκλήματος, ιδίω όταν ε, μπορούν να δημιουργηθούν μεγάλα κέρδη για αυτό το οργανωμένο έγκλημα. Δεύτερη κατηγορία, κυβερνοέγκλημα το οποίο οδηγεί σε σοβαρές βλάβες στα θύματα του και ένα από τα <clears throat> παραδείγματα είναι η σεξουαλική εκμετάλλευση στο διαδίκτυο και εδώ φυσικά υπήρξαν πολλές πολιτικές πρωτοβουλίες τέλος και μία ε, οδηγία για την σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών. Αυτό ήταν μια μεγάλη επιτυχία του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που συμφώνησαν να έχουν ένα από τα πρώτα τέτοια εργαλεία για τον κυβερνόχωρο μετά από την έγκριση της συνθήκης της Λισαβόνας. Και τέλος, η τρίτη κατηγορία, τα είδη κυβερνοεγκλήματος που είναι πολύ σοβαρά γιατί πλήττουν κρίσιμες υποδομές, όχι μόνο υποδομές πληροφορίας αλλά γενικά κρίσιμες υποδομές εν γέννη. Η ανακοίνωση της Κομισιόν παρουσιάζει τις κύριες λειτουργίες αυτού του κέντρου για το κύβερνο έγκλημα. Η βασική ιδέα για αυτό το κέντρο είναι ότι θα πρέπει να δίδει τη δυνατότητα συγκέντρωση στοιχείων και του να είναι ένα, σημείο, ένα εστιακό σημείο για την συσσόρευση ε, πληροφοριών. Σήμερα αυτό γίνεται σε επίπεδο Europol, αλλά θα έρθω μετά στο θέμα της εγκατάσταση αυτού του κέντρου. Έχουμε αυτή τη στιγμή στοιχεία από τις διοκτικές υπηρεσίες, αλλά ο στόχος μας στο μέλλον είναι να υπάρχει και ανάλυση πληροφοριών που έρχεται και από τον ιδιωτικό τομέα, από ανοιχτέ πηγές, από ερευνητές και από άλλους, άλλες χώρες κτλ. Ώστε έτσι το κέντρο αυτό να είναι καλύτερα προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει τους τρόπους με τους οποίους γίνεται το έγκλημα. θα έχει μεγαλύτερη δυνατότητα να δει νέους τρόπους με τους οποίους μεταλλάσσεται το κυβερνοέγκλημα. Δεύτερον, η ιδέα είναι... Η ιδέα είναι λοιπόν να προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε την εμπειρογνωμοσύνη που υπάρχει για το κυβέρνο έγκλημα που υπάρχει στα κράτη-μέλη και να υποστηρίξουμε ακριβώς την δυνατότητα ανάπτυξης αυτής της ε, αντίδρασης, μία από τις λειτουργίες του κέντρου αυτού θα ήταν ακριβώς να ε, ευθυγραμμίσει σε εισαγωγικά τις διαδικασίες ε, οι οποίες γίνονται και η μία να είναι συμπληρωματική της άλλης. Ένας από τους βασικούς στόχους θα είναι η δυνατότητα να υπάρξουν ad hoc συμβουλευτικές ικανότητες στα πλαίσια των υποθέσεων που οι ανακριτές ερευνητές αντιμετωπίζουν. Τρίτη λειτουργία είναι βασικό χαρακτηριστικό της Europol, το κάνει η Europol σήμερα, είναι να έρθει αρρωγό στα κράτη-μέλη σε επίπεδο ανακρίσεων, ερευνών. Νομίζουμε ότι η επένδυση αυτή, η οποία πρέπει να γίνει στο κέντρο αυτό για το κυβέρνο έγκλημα, η ποιότητα των, του ανθρώπινου δυναμικού θα αυξηθεί, θα βελτιωθεί και η κοινότητα αυτών των ερευνητών του κυβερνοχώρου μέσω του κέντρου θα έχει έναν μεγαλύτερο χώρο και θα ακουστεί συλλογικά στις αρχές επιβολής της τάξης και νόμου και θα είναι μια ουσιαστική πλατφόρμα για την διαδραστική επικοινωνία με τον ιδιωτικό χώρο αλλά και με τα κοινοτικά όργανα και με αυτούς οι οποίοι λαμβάνουν αποφάσεις. Τώρα για το πού θα είναι το κέντρο αυτό, αυτό ήταν ένα από τα βασικά προβλήματα τα οποία αναλύσαμε. Αρχικά, ξέρετε, ακούστηκαν πάρα πολλά σενάρια για το πού θα μπορούσε να είναι ένα τέτοιο κέντρο. Ίσως κάποιο κράτος μέλος το οποίο θα μπορούσε να αναλάβει μια τέτοια λειτουργία και για τα άλλα κράτη-μέλη. ένα θα έλεγα Έγιναν λοιπόν κάποιες συζητήσεις, έγιναν κάποιες προτάσεις για να υπάρξει ένα κέντρο στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών δομών. Προφανώς εμείς προσπαθούμε να είμαστε σε επαφή με τις κοινότητες, τις κοινότητες, αλλά Παρά όλα αυτά, το θέμα είναι να υπάρξει άμεση ανταπόκριση σε προβλήματα ε, διάπραξης εγκλημάτων, σε αποτελεσματικότητα ε, στη δίωξη των ε, εγκληματιών και αυτά όλα εντάσσονται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Europol και η Europol πράγματι έχει κάνει αρκετές έρευνες τον τελευταίο καιρό για την ανάπτυξη αυτής της δυνατότητας. Αυτή η επιλογή λοιπόν ήταν μια λογική επιλογή και σε επίπεδο λιτότητας επειδή δεν υπάρχει μεγάλη διάθεση για τη δημιουργία νέων κέντρων και νέων υπηρεσιών. Έχοντας πάρει την απόφαση λοιπόν να φιλοξενηθεί το κέντρο αυτό στο εσωτερικό της Αεροπόλ, έχει υπάρξει μια πολύ σημαντική πρόταση καινοτομική να υπάρξει δηλαδή ένας προγραμματικός πίνακας, ένα πλαίσιο προγραμματικό το οποίο να συλλέγει και να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις όλων των εμπλεκομένων οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με την ανταπόκριση στα κυβερνοεγκλήματα αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες συνδεσμολογίας που πρέπει να υπάρχουν. Η Eurojust θα συμμετέχει, η ENISA, η SIPOL, η ΣΥΠΟΛ μάλλον, που είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση των αστυνομικών. Τα κράτη-μέλη θα εκπροσωπούνται επίσης μέσω μιας υπάρχουσας μη επίσημης δομής της ε, ομάδας δράσης UCTF, όπου υπάρχουν τα λεγόμενα κόψε εκπρόσωποι του Συμβουλίου, στο Συμβουλίο των Κρατών Μελών και συναντώνται και ανταλλάσσουν πληροφορίες. Είναι κάτι το οποίο εδώ και δύο χρόνια λειτουργεί. Και την Ιουσέρτ η μαλλον μια μοναδα έχει σαν βασικό ρόλο να διασφαλίσει την ασφάλεια σε επίπεδο ε, κυβερνοχώρου των ευρωπαϊκών υπηρεσιών. Στόχος λοιπόν αυτού του προγραμματικού πλαισίου είναι να δίδει τις κατάλληλες συμβουλές, να μην παρεμβαίνει φυσικά στις κανονικές τακτικές διαχειριστικές δομές της Ευρωπόλ, όπου υπάρχει το Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο εκπροσωπούνται τα κράτη-μέλη. Το θέμα των πόρων, το δημοσιονομικό, αυτό ήταν ένα από τα πιο δύσκολα θέματα τα οποία είχαμε να αντιμετωπίσουμε προετοιμάζοντας αυτήν την ανακοίνωση. Είναι σαφές ότι ο χρονισμός δεν είναι ο κατάλληλος, βιώνουμε περιόδους λιτότητας, συζητήσεις για οριζόντιες μειώσεις, για την δυνατότητα μείωσης γενικότερα του κόστους και στις εξωτερικές υπηρεσίες και οι συζητήσεις που γίνονται οι διαπραγματεύσεις για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, πολιετές Οπότε δεν μπορούσαμε σε ένα τέτοιο πλαίσιο εμείς να επιδιώξουμε να κάνουμε δηλώσεις για τις νέους πόρους που θα απαιτούσε ένα τέτοιο κέντρο. Γι' αυτό και η ανακοίνωση αναφέρεται σε περαιτέρω αξιολογήσεις και υπολογισμούς που θα πρέπει να γίνουν πριν το κέντρο αυτό πράγματι λειτουργήσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου και εδώ υπολογίζουμε και στη δική σας βοήθεια όταν έλθουμε στη συζήτηση των δημοσιονομικών. Και σε επίπεδο βραχυπρόθεσμο και σε επίπεδο του πολιετούς ε, δημοσιονομικού προγραμματισμού. Έγινε μια μελέτη εφικτότητα σε εισαγωγικά η οποία έχει δημοσιοποιηθεί και η οποία, και δίνει μια ιδέα για τα ποσά τα οποία μπορεί να απαιτηθούν και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ε, δαπανηθούν. Είναι μια πρώτη εικόνα βέβαια, δεν είναι μια πλήρης απάντηση σε σχετικά, σχετικά με το επίπεδο των πόρων. Πάντως ε, εκφράζονται κάποιες βασικές ιδέες, κάποιες θέσεις οι οποίες θα μπορούσαν να απροστεθούν στις αντίστοιχες δραστηριότητες για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος της Ευρωπόλ. Θα είναι επίσης και μια πλατφόρμα διεθνούς συνεργασίας. Πολλά συμβαίνουν σήμερα στον κόσμο γύρω από αυτό. Μία από τις πρωτοβουλίες τις οποίες λαμβάνουμε υπόψη μας είναι το σχέδιο για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου ευρωπαϊκού κέντρου της Interpol στη Σιγκαπούρη και το Ευρωπαϊκό Κέντρο θα είναι στο πλαίσιο αυτό μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή συνεισφορά. Βασική ιδέα είναι φέτος να ξεκινήσουμε την εφαρμοστική φάση. Η ομάδα να αρχίσει να εργάζεται στο εσωτερικό της Ευρωπόλ το θέμα της ε, ουσιαστικής εμπλοκής όλων των συμμετεχόντων και της πρόκλησης ενδιαφέροντος είναι κάτι το οποίο θα τονιστεί κυρίως του χρόνου όταν ξεκινήσει η πραγματική λειτουργία και θα πρέπει ήδη από τις αρχές της λειτουργίας και τα, όλα τα κράτη-μέλη να μπορούν να συμμετέχουν και να επηρεάσουν τις εξελίξεις και στόχος μας είναι το 2013 το κέντρο αυτό να ξεκινήσει τις δραστηριότητές του πάνω το συνολικό σύστημα και ο τρόπος με τον οποίο οι λειτουργίες θα φανούν αποτελεσματικές θα εξαρτηθούν από τους πόρους τους οποίους μπορούμε να διασφαλίσουμε και θα είστε και εσείς ικανοί να διασφαλίσετε. Τέλος, πολλά ζητούνται από τα κράτη-μέλη σε σχέση με τις δυνατότητες τις οποίες έχουν σε επίπεδο διεθνούς συνεργασίας για να μπορέσουν όλοι να προσφέρουν στο κέντρο αυτό. Είχαμε πολλές απαντήσεις από τα κράτη-μέλη Ξέρετε ότι ε, το ζήτημα αυτό το συζητάμε τώρα και θέλουμε κατά τη διάρκεια της Δανέζικης Προεδρίας να έχουμε συμπεράσματα του Συμβουλίου υπέρ της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου για Κλίματα στον κυβερνοχώρο που θα πρέπει να εγκριθούν μέχρι τα τέλη του έτους. Έχουμε πάντως ένα σημαντικό ενδιαφέρον και σημαντική υποστήριξη από πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παράλληλα, διεξάγονται και διαπραγματεύσεις για την ε, οδηγία για τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Η Επιτροπή ε, Πολιτικών Ελευθεριών ασχολείται με, την, ε, με το ζήτημα αυτό και έχουμε και την υποστήριξη λοιπόν των Ευρωβουλευτών και προσβλέπουμε βέβαια να συνεχιστεί η υποστήριξη αυτή κατά τη διάρκεια της θέσπισης και της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα Εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, ιδίως ε, εφόσον δεν έχει λυθεί ακόμα το ζήτημα των πόρων της χρηματοδότησης. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που μου δώσετε την δυνατότητα να σας παρουσιάσω τα σημαντικότερα δεδομένα όσον αφορά την δημιουργία του κέντρου αυτού. Θα θέλαμε βέβαια και κάποια στιγμή στο μέλλον να είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε για το πού θα έχουμε φτάσει τότε. και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρωτοβουλία αυτή είναι πολύ σημαντική και πιστεύουμε ότι μπορεί να συμβάλλει πολύ σημαντικά στην αντιμετώπιση όλων αυτών των απειλών στα πλαίσια του κυβερνοχώρου. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Μία ερώτηση θα ήθελα να θέσω. Για μένα οι επιθέσεις του κυβερνοχώρο δεν είναι μόνο εγκλήματα στον κυβερνοχώρο έχουν να κάνουν και με την στρατιωτική κατάσταση κάθε φορά. Από όσο κατάλαβα, εσείς δεν έχετε καμία στρατιωτική προσέγγιση στην πρωτοβουλία σας. Αναφέρεστε μόνο για τα, στα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο. Επίσης, χρειαζόμαστε μια κοινή νομική υποστήριξη για τη δραστηριότητα αυτή. Όταν λέτε ότι θέλετε να συγκεντρώσετε εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναφέρεστε σε αυτά τα οποία ήδη γνωρίζουν τα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων. Η κυρία Κοπά το λόγο. Θα λάβω το λόγο εξ ονόματος του κυρίου Γιάννης Μπαριονουέβο που δεν μπόρεσε να είναι παρόν. Τα σχόλιά του για την έκθεση είναι τα εξή. Λέει καταρχήν είναι πράγματι γεγονό ότι γίνεται μια παγκόσμια πρόκληση για την κοινωνία μα το κυβερνό έγκλημα και οι Ευρωπαίοι πολίτε έχουν όλο και μεγαλύτερη επίγνωση ανάγκη να αυξήσουν την κυβερνοασφάλεια. Είδαμε μεγάλο ενδιαφέρον την ανακοίνωση τη Κομισιόν και θα ήθελα να πω ότι χαιρετίζω την πρόταση να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο για το έγκλημα, που είναι μια διαμεθοριακή απειλή και γι' αυτό πιστεύω ότι χρειάζεται συντονισμένη δράση που να συμπεριλαμβάνει και τι εξωτερικέ πολιτικέ ασφάλειες. Αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κυβέρνο Εγκλήματος θα πρέπει να συμπληρωθεί, με ένα πιο εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο και περισσότερους πόρους σε επίπεδο κρατών μελών. Και επίσης πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την διαμόρφωση και τον έλεγχο αυτού του κέντρου. Αυτά λέει ο κ. Μπαριονούεβο. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω εξ ονόματος της μου την ανάγκη η οποία αναφέρεται ήδη στα σχόλια του κ. Νουέβο του να υπάρξει ένα νομικό πλαίσιο, γιατί χωρίς νομικό πλαίσιο δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει τίποτα τέτοιο. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν ποια είναι η άποψή σας για τη δυνατότητα να έχουμε το απαραίτητο αυτό νομικό πλαίσιο. Κυρία Λούζινγκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και καυτό θέμα αυτό <clears throat> όταν πρόκειται για την εγκληματική κατάχρηση του διαδικτύου και αυτό είναι ένα πολύ ευρύ θέμα φυσικά. Πιστεύω ότι είναι θεμητό, θεμητή διεκδίκηση των πολιτών να εξασφαλίσουν την προστασία από αυτές τις εγκληματικές ενέργειες, αλλά υπάρχει και μία, ένα δικαίωμα των πολιτών να προστατευθούν τα πολιτικά και αστικά τους δικαιώματα και η έννοια της δημοκρατίας. Και εδώ υπάρχει μια ένταση μεταξύ των δύο αυτών διεκδικήσεων, των δύο αυτών μορφών δικαιωμάτων. Το ανέφερε και η πρόεδρος μας, η κυρία Νικολάη, όταν είπε ότι το θέμα αυτό έχει και μια στρατιωτική διάσταση και φυσικά βρισκόμαστε στην Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας. Εγώ ενοχλούμε προσωπικά για το γεγονός ότι η Κομισιόν κάπως αφήνει κατά μέρο τη στρατιωτική πτυχή του θέματος αυτού και έχω πολλές ανησυχίες ότι όλα αυτά τα θέματα θα μπουν από την πίσω πόρτα στο κέντρο αυτό. Στην ε, Γερμανία έχουμε ήδη ένα εθνικό κέντρο άμυνας εναντίον των επιθέσεων των hacker το οποίο έχει δημιουργηθεί και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δημιουργίας αυτού του κέντρου υπήρξαν πάρα πολλές συζητήσεις και διαμάχες σε σχέση με την διασύνδεση μυστικών υπηρεσιών με αστυνομία και στρατιωτικές υπηρεσίες κτλ. Και επομένως εδώ βρίσκεται η δική μου ανησυχία αν θα προκύψει και κάτι τέτοιο, γιατί όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλους κινδύνους για τη δημοκρατία και την διαφάνεια των διαδικασιών και την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω μέσα σε ποιο πλαίσιο θα δημιουργηθεί αυτό το κέντρο ευρωπαϊκού χαρακτήρα, πώς θα υπάρχει η ανταλλαγή απόψεων, θα γίνεται με τη συμμετοχή μυστικών υπηρεσιών και στρατιωτικών φορέων και όλα αυτά πώ θα συνδυαστούν με την ε, Europol. Αυτό μου φαίνεται κάπω δύσκολο να το, καταναήσω. Θα ήθελα λοιπόν να έχω περισσότερη διευκρίνηση για τα θέματα αυτά. Ίσως θα μπορούσατε να μου δώσετε εσεί περισσότερε εξηγήσει εκπρόσωπε τη Κομισιόν. Κύριε Κέλαμ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ενθαρρύνομαι από αυτή την πρωτοβουλία της Κομισιόν είναι πολύ καλά τεκμηριωμένη και εδρεωμένη. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε καταρχήν ότι θα πρέπει να προσβλέψουμε στην ε, πραγματοποίηση αυτής της ε, πρωτοβουλίας. Το ερώτημα μου είναι το εξής. Είπατε καταρχήν στην παρουσίασή σας ότι η κύρια βάση σε νομικό επίπεδο είναι η Σύμβαση της Βουδαπέστης για το κυβερνό έγκλημα, που είναι μια σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Θεωρείται όμως ότι επαρκεί αυτή η σύμβαση ως νομική βάση. <clears throat> Μήπως χρειάζεται κάποιο εξυγχρονισμό αυτή η σύμβαση ή κάποια διεύρυνση ή θεωρείτε ότι μπορείτε να καλυφθείτε στο άμεσο μέλλον από αυτήν την σύμβαση και μόνο. Επίσης η Κομισιόν αναφέρεται σε ορισμένα προσκόμματα για τη συνεργασία στα θέματα αυτά και αναφέρει παραδείγματος χάρη τα διαφορετικά νομικά συστήματα και το πώς δύσκολο να ξεπεράσει κανείς τα εθνικά σύνορα για τα θέματα αυτά. Έχετε και κάποια σχέδια για το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα, γιατί πράγματι είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Επίσης αναφερθήκατε και στην έλλειψη επαρκών μέσων για τον επιμερισμό των πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και <clears throat> μεταξύ των εμπλεκομένων. δείχνετε να είστε διστακτικός ή <clears throat> επιφυλακτικός σε σχέση με την αίτηση περαιτέρω για το κέντρο αυτό. Πώς θα ξεπεραστεί όμως το πρόβλημα αυτό της ανεπάρκειας των πόρων για την συλλογή και την ε, θέση από κοινού των πληροφοριών. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό ερώτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε, γιατί αυτό το κέντρο θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να τίθεται από κοινού η πληροφορία, αλλά οι πληροφορίες αυτές από την ίδια τη φύση τους είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες και εμπιστευτικές. Πώς θα γίνει κάτι τέτοιο, πώς παραδείγματος χάρη θα έχουν πρόσβαση εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα σε, αυτά τα, σε αυτές τις πληροφορίες. Αυτό είναι το ερώτημα που ήθελα να σας θέσω. Κύριε Γκάλερ, ευχαριστώ. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι με έχουν καλύψει γιατί έχουν θέσει όλα τα ενδιαφέροντα ερωτήματα. Εγώ έχω μονάχα ένα μικρό ερώτημα που αφορά τις ε, πολιτικές μας ε, αποστολές ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα... Πώς έχει γίνει μάλλον μέχρι τώρα η προστασία για την Κομισιόν των ε, συστημάτων υπολογιστών που υποστηρίζουν τέτοιου είδου αποστολέ. Τι έχει γίνει μέχρι τώρα, γιατί λέτε ότι πρέπει να υπάρχει μια κοινή δομή, αλλά τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, πώς λειτουργεί το σύστημα αυτή τη στιγμή για κοινέ αποστολέ. Ο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, θα πρέπει να διακρίνουμε διάφορες πτυχές στα πλαίσια της κυβερνοασφάλειας, των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο. Πτυχές που έχουν και πολιτικές και στρατιωτικές διαστάσεις. Και βέβαια πρέπει να μιλήσουμε συγκεκριμένα και για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο. Ούτως ή άλλως η ανακοίνωση αυτή σε αυτό εστιάζεται. Θα ήθελα να γνωρίζω αν τελικά αυτό το οποίο προτείνεται είναι να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο ή απλώς να δημιουργήσουμε ένα ακόμα όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε ότι το πρόβλημα αυτό είναι διεθνές. Πολλά από τα εγκλήματα αυτά ουσιαστικά προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να εστιαστούμε και στην εξωτερική αυτή διάσταση και θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή και με άλλες, και με άλλες χώρες και με άλλους οργανισμούς και δεν ξέρω ποιες θα είναι οι επιπτώσεις όσον αφορά τους σπόρους τις δαπάνες. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία της ανακοίνωσης, ενώ τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφιερώνει μια πολύ μικρή παράγραφο. Αναφέρομαι στις δαπάνες. Πώς θα κοστίσει το εγχείρημα, από πού θα έρθουν οι πόροι. Αν πρόκειται για κοινοτική αρμοδιότητα, τότε τι περικοπές θα γίνουν σε άλλους τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να βρεθούν οι απαραίτητοι πόροι για να λειτουργήσει, να στηθεί αυτό το Ευρωπαϊκό Κέντρο το οποίο προτείνεται. Νομίζω ότι τα ερωτήματα αυτά είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να απαντηθούν. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε κύριο Σάρενχάουζερ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να εφερθώ στο ζήτημα των πόρων. Από ό,τι φαίνεται, υπάρχει κάποιο όριο, μέχρι το οποίο μάλλον βάσει το οποίο μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την όλη πρωτοβουλία θετική ή αρνητική. Πρέπει να δούμε για παράδειγμα το προσωπικό, πόσοι άνθρωποι θα απασχοληθούν, αν θα δημιουργηθεί κάποιο γραφειοκρατικό άκθος από τον νέο αυτοοργανισμό ή όχι. Εσείς είπατε ότι έχετε ήδη ένα διαθέσιμο προσωπικό έχετε αποφασίσει κάποια πράγματα για την έδρα, αλλά τι πόρους τελικά θα χρησιμοποιήσουμε για το κέντρο αυτό και αν τελικά αποτελέσει μέρος της Europol θα εξαρτάται και από τον προπολογισμό της Europol και αν ισχύει κάτι τέτοιο τότε θα απορροφηθεί προσωπικό της Europol ή τα πράγματα θα κινηθούν εντελώ διαφορετικά για αυτόν τον οργανισμό θα μπορούσαμε να προβλέψουμε μια κάποια συγχώνευση. Για παράδειγμα, έχουμε και την ΕΝΙΣΑ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών και δεν νομίζω ότι έχει επιλεγεί καλύτερη δυνατή έδρα για την ΕΝΗΣΑ. Θα μπορούσαμε να συγχωνεύσουμε την ΕΝΙΣΑ με ένα τέτοιο κέντρο ή αν αυτό θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε κάποιες εξοικονομήσεις πόρων. Ένα ακόμα περαιτέρω ερώτημα για του στόχου της δημιουργίας ικανότητα στα κράτη-μέλη για την ασφάλεια των υπηρεσιών. Μπορείτε να μας πείτε πώς θα μπορέσετε με τον τρόπο αυτό να αντιμετωπίσετε την ικανότητα των κρατών μελών και ποιες είναι οι τωρινές ικανότητες αυτών των κρατών μελών, πώς θα μπορούσε να γίνει μια συλλογική ε, συγκέντρωση όλων αυτών των μέσων όταν έχουμε την προστασία των παιδιών από το, την πορνογραφία και το έγκλημα, δεν νομίζω ότι οι τωρινέ ικανότητε που υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο θα μπορούσαν να επαρκέσουν για ένα τέτοιο στόχο. Αυτά ήθελα να πω. Έχετε το λόγο για να απαντήσετε για τα πολλαπλά αυτά ερωτήματα. Yeah, I try my best uh, to, at least to, to... Θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου για να απαντήσω κάποιες από τις ερωτήσεις, σε κάποιες από τις ερωτήσεις για τη στρατιωτική διάσταση. Αυτό δεν είναι κάτι που εξετάζουμε. Δεν είναι αρμοδιότητά μας, δεν υπάρχει τέτοια αρμοδιότητα, αλλά όπως είπατε τα θέματα αυτά συνδέονται. Και όταν υπάρξει μια περίπτωση κυβερνοεπίθεσης και εφόσον δεν γνωρίζουμε το ποιος την έχει διαπράξει ή οσδήποτε θα μπορεί να κρύβεται από πίσω. Είτε ένας εγκληματίας, είτε μια τρομοκρατική ομάδα, είτε μια χώρα. Obviously this is beyond the remit of, Center. Πάντως αυτό το κέντρο θα συγκεντρώσει την προσοχή του στις ποινικέ πλευρές. Θα προσπαθήσει να, να εντοπίζει δηλαδή αυτούς οι οποίοι ε, διαπράττουν τις επιθέσεις και να αναζητεί τους τρόπους να τους κατηγορήσει επίσημα. Σχετικά με την εμπειρογνωμοσύνη, αναφερόμαστε πιο συγκεκριμένα σε γνώσεις για νέου τύπου επιθετικά, επιθετικούς ιούς που χρησιμοποιούνται για την διάπραξη υποκλοπής στοιχείων, phishing ή α, κυβερνοεπιθέσεων επίσης ε, γνώση ε, της λειτουργίας ε, εγκληματικών ενεργειών που διευκολύνονται μέσα από το διαδίκτυο όπως πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς χρήσης ταυτοτήτων άλλων υπολογιστών για τη διάπραξη επιθέσεων που δημιουργούν προβλήματα, μπλοκάρουν ιστοσελίδες Γνωρίζουμε ότι κάποιοι άλλοι υπολογιστές χρησιμοποιούνται επίσης και για εκβιασμούς. Λοιπόν, θα μπορούσα να δώσω και άλλα παραδείγματα, ένα μόνο, για το ρόλο του κέντρου σε επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης, θα είναι η συλλογή και επεξεργασία ιατροδικαστικών μέσων, δηλαδή και λογισμικών και ίσως κάποιων ε, εξοπλισμών ηλεκτρονικών για την ανάλυση σκληρών δίσκων, άλλων υπολογιστών, για την ανάλυση ε, υπόπτων ε, λογισμικών κτλ. Για όλα αυτά λοιπόν σωστά υπόθηκε ότι το βασικό νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμε θα είναι η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης της Βουδαπέστης για το κυβέρνο έγκλημα παρότι έγινε δεκτή σύμβαση αυτή το 2001, λόγω του τρόπου με τον οποίο έχει συνταχθεί και λόγω των, θα έλεγα, σκοπιμοτήτων αυτών που το συνέταξαν, είναι τεχνολογικά ιδέτε, ουδέτερο και γι' αυτό ακριβώς επιτρέπει τον σωστό εντοπισμό των μέσων που είναι απαραίτητα για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος και επιτρέπει επίσης και τη δικαστική συνεργασία. Η σύμβαση λοιπόν αυτή του Συμβουλίου της Ευρώπης επιτρέπει την δημιουργία νέων και εκτιμένων, προστατεύει τα συστήματα πληροφόρησης από τις κυβερνοεπιθέσεις και αναθεωρούμε το νομικό μέσο που έχουμε εμεί στη διάθεσή μας και έχουμε τη συζήτηση για την οδηγία για τις κυβερνοεπιθέσεις η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε λίγο πέραν της συμβάσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης. This is a part of European legislation, unlike in the Council of Europe Convention. Uh, Σχετικά με τα ρομποτικά, τα botnets, τα ρομποτικά προγράμματα, να προχωρήσουμε στην δυνατότητα επιβολής ενός ελαχίστου επίπεδου ποινών όταν κάτι τέτοιο χρειάζεται. Τώρα για τις πιθανές ανησυχίες που υπάρχουν για τις επιπτώσεις για τους ε, πολίτες και για τις δραστηριότητες των πολιτών σχετικά με την προστασία τους από το κυβέρνο έγκλημα. Να πω ότι το πλεονέκτημα του να υπάρχει κάτι τέτοιο στο εσωτερικό της Ευρωπόλη είναι ότι στα πλαίσια της Ευρωπόλη έχουμε ισχυρότατα συστήματα ελέγχου και προστασίας των προσωπικών δεδομένων για την ανταλλαγή ε, πληροφοριών και την δυνατότητα ανάλυσης και εξέτασης φακέλων. Αυτό μας δίνει, θα έλεγα, την πεποίθηση, μας δημιουργεί την πεποίθηση ότι έχουμε στη διάθεσή μας υψηλά επίπεδα προστασίας που είναι απαραίτητα τελικά για την πρόληψη καταχρήσεων. Ίσως δεν θα έπρεπε να απευθύνω μια τέτοια πρόκληση από πλευρά τη Ευρωπόλ, αλλά ξέρω ότι η Ευρωπόλ ήδη έχει ε, φιλοξενήσει τον κύριο Χολμάγερ, ο οποίος είναι ο εισηγητής για τα θε... την κυρία Χολμάγερ, η οποία είναι η εισηγήτρια, για τα θέματα της προστασίας από επιθέσεις στο κέντρο της. Ίσως ξέρετε ότι αυτός, πιστεύω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να συλλάβετε πραγματικά την ποιότητα της εργασίας η οποία έχει ήδη γίνει και θα γίνει στο μέλλον στα πλαίσια αυτού του κέντρου. Yes, question of private sector. Uh, of Το θέμα είναι να υπάρξει και ένα άνοιγμα του κέντρου και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Θα πρέπει όμως να κάνουμε μια διάκριση εδώ ανάμεσα στα είδη της πληροφόρησης και της ανταλλαγής πληροφοριών που μπορεί να υπάρξει. Όταν έχουμε να ανταλλάξουμε πληροφορίες για έρευνες, για υπόπτους, αποδείξεις, ανακριτικές διαδικασίες, όλα αυτά μπορεί να ανταλλαγούν μόνον, μόνον με έναν πολύ προστατευμένο, αυστηρά προστατευμένο τρόπο ανταλλαγής πληροφοριών, ο οποίος ισχύει αυστηρά για τις δυνάμεις καταστολής και επιβολής τάξης. Όταν μιλάμε για ανταλλαγή πληροφοριών με τον ιδιωτικό τομέα, το θέμα είναι ο ιδιωτικός τομέας να μας ενημερώνει για νέους τρόπους τέλεσης κυβερνοεπιθέσεων, για νέα τεχνολογικά μέσα καταπολέμησης ε, του κυβερνοεγκλήματος, για τον εντοπισμό νέων μορφών επιθετικών ιών, Υπάρχει εδώ σημαντικό πεδίο θα έλεγα το οποίο ξεπερνά το θέμα μόνο του κέντρου αλλά υπάρχει ένα διαφορετικό πρόβλημα αντιμετώπισης του κυβερνοεκκλήματος σήμερα και αυτό οφείλεται στο ότι οι περισσότερες από τις κυβερνοεπιθέσεις ποτέ δεν ανακοινώνονται στις δυνάμεις καταστολής. Ε, γιατί γίνεται αυτό, κοιτάξτε, πολλές φορές μιλάμε για πιστοτικά ιδρύματα, τα οποία για προφανείς λόγους, λόγους εμπιστοσύνης, δεν θέλουν να δώσουν αυτή την ενημέρωση και οι αρχικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως και των τροπολογιών του Κοινοβουλίου στην ε, οδηγία η οποία είναι υποδιαπραγμάτευση δημιουργείται μια κάποια μορφή υποχρέωσης δημοσιοποίησης των επιθέσεων και των θυμάτων. Είναι κάτι το οποίο αυτό δεν αναφέρεται άμεσα στο κέντρο βέβαια, γιατί αυτές οι υποχρεώσεις αναφέρονται σε επίπεδο δημοσιοποίησης ε, ανακοίνωσης των επιθέσεων σε εθνικό επίπεδο αλλά η εικόνα η καλύτερη που θα έχουμε για τις επιθέσεις οι οποίες διαπράττονται δεν θα βοηθήσουν μόνο γενικά τις προσπάθειές μας, αλλά θα βελτιώσουν την δυνατότητα αντιμετώπισης του σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εφόσον οι πληροφορίες αυτές μεταφερθούν στην Ευρωπόλ από τις εθνικές αρχές, αστυνομικές αρχές. Σας ευχαριστώ για τις ανησυχίες τις οποίες εκφράσατε και εσείς για τους πόρους. Νομίζω ότι ήμουν αρκετά δεκτικός λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι εν γνώση του τι θα θέλατε να περιλαμβάνει μια τέτοια ανακοίνωση, πιο ξεκάθαρα στοιχεία. Αλλά από την άλλη σας εξήγησα και για ποιο λόγο δεν ήταν δυνατόν να έχουμε αυτά τα ξεκάθαρα στοιχεία, γιατί δεν έχει υπάρξει μια συμφωνία η δυνατότητα, η μελέτη εφικτότητα σε εισαγωγικά δίνει κάποιες πρώτες ιδέες για το κόστος αυτό. Είχε προτείνει σαν παράδειγμα έναν προϋπολογισμό της Ευρωπόλ να αυξηθεί κατά 3,5 περίπου εκατομμύρια το 2013 και συνολικά όταν λειτουργεί πλήρως το κέντρο να φτάσουμε σε επιπλέον 8 εκατομμύρια. Αυτή είναι μια πρώτη ιδέα του βάρους του οικονομικού που θα δημιουργηθεί στις συγκεκριμένες θέσεις του προϋπολογισμού από το 2013 ή 2014. Ελπίζω να μην κάνω λάθη εδώ, αλλά όλα αυτά θα μπορέσετε να τα βρείτε στη μελέτη. Πάντως ε, θα έλεγα είναι μία πρώτη μελέτη. Αυτή σε καμία περίπτωση δεν είναι μία υποχρέωση την οποία αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως σας είπα δίνει όμως κάποιες πρώτες ε, ε, εικόνες τεχνικά τα θέματα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τον προϋπολογισμό της Ευρωπόλ. Μιας και το κέντρο αυτό θα, θα, θα, λειτουργήσει στο εσωτερικό των δομών της Ευρωπόλ, πρέπει να καλυφθεί δημοσιονομικά από την Ευρωπόλ. Αυτό θα αντικατοπτρίζεται και στο, στον προϋπολογισμό της Ευρωπόλ και στο ανθρώπινο δυναμικό στο οργανόγραμμα της Ευρωπόλ είναι κάτι το οποίο έτσι και αλλιώ θα πρέπει να αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου ε, λογαριασμού, ενός ευρύτερου πλαισίου. Για την προστασία των συστημάτων των ηλεκτρονικών που χρησιμοποιούνται στις εξωτερικές δράσεις, αυτό δεν μπορώ να δώσω απάντηση. Δεν ασχολούμεθα με τις εξωτερικές πλευρές τέτοιου είδους δράσεων αυτό δεν είναι τμήμα των αρμοδιοτήτων της δικής μου υπηρεσίας. Πάντως νομίζω ότι το θέμα αυτό μπορώ να το μεταφέρω και να πάρετε κάποιες απαντήσεις. Σχετικά με την ενίσα. Εδώ είναι αρκετά διαφορετικές οι εντολές των δύο φορέων. Ο ρόλος της ενίσα είναι να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να αυξήσουν την ανθεκτικότητα των συστημάτων πληροφόρησης τους, να υποστηρίξουν προληπτικές γενικά ενέργειες εναντίον ενός ευραίως φάσματος κύβερναπηλών και βέβαια δεν χρειάζεται να είναι απειλές οι οποίες είναι ανθρωπογενείς όπως συμβαίνει στην περίπτωση του κυβερνοεγκλήματος. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μία προφανής συνέργεια γιατί η κυβερνοασφάλεια συμβάλλει στην πρόληψη, πιο ανθεκτικά συστήματα ασφαλείας είναι πιο δύσκολα για τους ε, εγκληματίες του κυβερνοχώρου να διεισδύσουν σε αυτά. Αν οι τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της χάρη, προωθήσουν το σύστημα των ε, tokens όταν ε, συνδέεται κανείς ηλεκτρονικά με την τράπεζά του ε, κανείς. Με τον τρόπο αυτό υπάρχουν λιγότερες περιπτώσεις phishing, δηλαδή παράνομης απόκτησης των, ε, της ταυτότητας του χρήστη. Επομένως είναι συνδεδεμένα αυτά τα θέματα. Η Ενίσα θα λαμβάνει μέρος στο Συμβούλιο του νέου αυτού κέντρου και θέλουμε στο κέντρο αυτό διάφοροι εμπλεκόμενοι όπως η EU CERT και η ENISA να μπορούν να <clears throat> αποσπούν προσωπικό στη Χάγη σε μόνιμη βάση, ώστε να υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι ο σύνδεσμος των κέντρων αυτών, των φορέων αυτών με το κέντρο και εξασφαλίζει έτσι ότι υπάρχει το αίσθημα της πλήρους συμμετοχής. Όλα αυτά φυσικά εξαρτώνται από τους διαθέσιμους πόρους, αλλά αυτή είναι η κατεύθυνση στην οποία θέλουμε να κινηθούμε. Τέλος, υπήρχε ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα για το θέμα της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στο διεθνές πλαίσιο. Αυτό είναι θέμα της ΙΠΑ ε, του εκπροσώπου. Αλλά για να σας πω ποια είναι η δική μας σκέψη για τα θέματα αυτά, γενικά η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι θεωρούμε ότι το τωρινό μοντέλο διακυβέρνησης που είναι διακυβέρνηση του διαδικτύου που δεν γίνεται από, το Ενωμένο, από τα ενωμένα Έθνη από άλλο φορέα δημόσιο αλλά η τωρινή διακυβέρνηση του ίντερνετ που γίνεται από ένα ιδιωτικό φορέα με μεγάλη συμμετοχή πολλών εμπλεκομένων <clears throat> υπάρχει γενικά μία συνένεση ότι για να εξασφαλίσουμε την ελευθερία και την δημιουργικότητα και την καινοτομία στο ίντερνετ πρέπει να διατηρηθεί μια τέτοια μορφή διακυβέρνησης του διαδικτύου και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι εναντίον των απόψεων της Κίνας ή της Ρωσίας για τη διακυβέρνηση του ίντερνετ και στο συγκεκριμένο τομέα του, κυβερνο, του εγκλήματος στον κυβερνόχωρο εμείς υποστηρίζουμε ιδιαίτερα την σύμβαση της Βουδαπέστης και δεν είμαστε πεπισμένοι ότι υπάρχει ανάγκη να προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσει για ένα νέο νομικό πλαίσιο στην, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Αυτή είναι η γενική κατάσταση. Νομίζω ότι υπάρχει μια γενική αντίληψη η οποία αντανακλά αυτά που είπατε στην Επιτροπή σας. Υπάρχουν πολλές δυνατές απειλές, υπάρχουν συνδυασμοί θεμάτων και προβλημάτων που μπορεί να άπτονται και της στρατιωτικής διάστασης. Η κάθε χώρα λοιπόν θα πρέπει να διατηρήσει ένα διάλογο για το πώς τα θέματα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, με τι τρόπο μπορούμε να έχουμε μέτρα υποστη... Ε, δημιουργίας εμπιστοσύνης χωρίς να αναπτύξουμε νέα διεθνή εργαλεία γιατί αυτό είναι ίσως κάπως δύσκολο. Μπορεί να γνωρίζετε ότι πρόσφατα έγινε μια συνδιάσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο πέρσι, όπου ο στόχος ήταν να συζητηθούν τα θέματα κανόνων συμπεριφοράς στο, στο κυβερνόχωρο. Υπήρξε εκπροσώπηση της Κομισιόν με την Επίτροπο κυρία Κρούζ, υπήρξαν εκπρόσωποι και 100 μελών και η ιδέα αυτή ότι πρέπει να συζητήσουμε περισσότερο και με τους Ρώσους και τους Κινέζους για ελάχιστες προδιαγραφές και πρότυπα σε σχέση με την δράση των κυβερνήσεων στο ίντερνετ. Είναι μια διαδικασία που θα συνεχίσει να εκτιλήσεται και όπου θα τεθούν πολλά τέτοια ερωτήματα και στο μέλλον. Η συνδιάσκεψη συνέχειας του Ηνωμένου Βασιλείου θα γίνει στην Ουγγαρία και ξέρουμε ότι η Ουγγαρία και πάλι παίρνει την πρωτοβουλία να σκεφτεί για τα θέματα αυτά το αν θα προκύψει κάτι το απτό από όλα αυτά. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουν οι συναδελφοί μα στην υπηρεσία εξωτερική δράση. Απλώ σα τα λέω για να ξέρετε ότι μια διαδικασία προβληματισμού είναι εν εξελίξη. Όλων και περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναπτύξει τη δική τη θέση για τα ζητήματα αυτά. Ελπίζω ότι έχω προσπαθήσει τουλάχιστον να απαντήσω τα περισσότερα ερωτήματά σας. Πολλές από τις απαντήσεις όμως θα μπορέσουμε να σας τις δώσουμε όταν έχει προχωρήσει η διαδικασία εγκαθίδρυσης αυτού του κέντρου και θα μπορέσουμε να επικαιροποιήσουμε τις πληροφορίες που σας δίνουμε. Ευχαριστώ. Άλλα ερωτήματα. Ένα τελευταίο ερώτημα. Ξέρετε ότι το ΝΑΤΟ έχει στην Ταλίν ένα κέντρο αριστείας θα συνεργαστείτε με αυτό το κέντρο για να συνενώσετε την εμπειρογνωμοσύνη σας παρά το γεγονός ότι είναι κάπως διαφορετική η τομή δράση, αλλά η εμπειρία αυτού του κέντρου μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη για να αντιμετωπιστεί το οργανωμένο έγκλημα. Υπήρξαν άτυπες συζητήσεις μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, στην οποία λάβαμε μέρος και εμείς και συμπεριλάμβανε αυτό, αυτή η συζήτηση τα συστήματα που έχει αναπτύξει το κέντρο της Σταλίν. Αλλά καταρχήν θεωρούμε ότι στην τρέχουσα χρονική στιγμή οι περισσότερες δραστηριότητες του ΝΑΤΟ αφορούν αποκλειστικά την προστασία της υποδομής σε πληροφοριακό επίπεδο του ΝΑΤΟ και των επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ. Ξέρουμε λοιπόν ότι οι συνάδελφοί μας από τις <clears throat> στρατιωτικές δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διάλογο με το ΝΑΤΟ, αλλά από ό,τι γνωρίζω δεν υπάρχει τίποτα το συγκεκριμένο που έχει προκύψει. Κοιτάξτε, στο Τάλιν της Εστονίας έχουμε και ένα κέντρο αριστείας το οποίο το υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ασχολείται με το ζήτημα της καταπολέμησης των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο. Επομένως και εκεί και σε αυτό το κέντρο έχουμε όλο και περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταθέτουν σχετικές πρωτοβουλίες. Υπάρχει ουσιαστικά ένα άτυπο δίκτυο κέντρων που συγκεντρώνουν πληροφορίες που έρχονται από κράτη-μέλη, από διάφορες επιστημονικές κοινότητες. Έχουμε τέσσερα κέντρα στην Ιρλανδία, τη Γαλλία, το Βέλγιο και την Εστονία. Και θα προκύψουν και άλλα κέντρα τα οποία θα κάνουν αίτηση χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε. Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Να σας ευχαριστήσω για την παρέμβασή σας, για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώσαμε και το δεύτερο σημείο στη μερίσια διάταξη σας προτείνω να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα προτού ξεκινήσουμε τη, συνεδρίαση του Διευρυθέντος Προεδρίου. Θα συνεχίσουμε και αύριο τη συνεδρίασή μας. Θα ξεκινήσουμε στις 9.30 το πρωί, στην ίδια αίθουσα νομίζω.